Κυρίε er gesagt? Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Sitzung Κυρίες και κύριοι, ξαναρχίζει η συνεδρίαση. Τα πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης σας διανεμήθηκαν. Δεν ξέρω κατά πόσο έχετε αντιρρήσεις επ' αυτών. Από ό,τι βλέπω όχι. Ε, κατόπιν τούτου ε, εγκρίνονται τα πρακτικά. Σύμφωνα λοιπόν με την ημερήσια διάταξη θα έχουμε τις δηλώσεις ε, του Συμβουλίου και της Κομισιόν για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τη Γάζα. Έχουμε την ιδιαίτερη χαρά ε, να μπορούμε να καλωσορίσουμε εδώ τον Υπουργό Εξωτερικών της Τσεχίας, ε, τον κύριο Σβάτσενμπεργκ, ο οποίος σήμερα το βράδυ θα πάει στη Νότια Αφρική και οι ε, παλαιότερες ε, προεδρίες έκαναν το εξής. Δεν ερχόντουσαν οι ίδιοι Υπουργοί Εξωτερικών, έστελαν τους αντικαταστάτες τους. Γι' αυτό ε, σας ευχαριστούμε θερμά κύριε Σφάτσενμπερκ για το γεγονός ότι ήρθατε σήμερα εδώ. Έχουμε και την κυρία Μπενίτα Φεραίρο Βάλτινα, την αρμόδια επίτροπο, η οποία επίσης γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα της Μέσης Ανατολής και η ίδια έχει ήδη πάει επί τόπου, όπως και ο κύριος Σφάτσεμπερκ. Αγαπητοί συνάδελφοι, λίγοι είμαστε εδώ, λίγοι αλλά καλοί. Ε,